Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι και ένας ίδιος πόρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you for your speech. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, το λόγο έχει ο συνάδελφος Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.